Οι ε, αρχές της ε, Λιθουανίας μας ανακοίνωσαν άρση της ε, ασυλίας του κυρίου Βίκτου Ουσπάτσης και σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού αυτό παραπέμπεται στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.